Ψηφιτητική εδώ πέρα μέσα το κοινοβούλιο. Ερχόμαστε να ψηφίσουμε και μας κατακλείζουν διάφοροι που θα μας δίνουν χαρτιά και φυλάδια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπράτμπερν για την ε, πρόταση αυτή που κάνατε, την οποία και θα ανακοινώσουμε, θα μεταβιβάσουμε στους ε, κοσμήτορες ε, έτσι ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Θα τις διαβάσω. Η αρμόδια επιτροπή έστειλε την διόρθωση ενός κειμένου το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίζει τις εναρμονισμένες προϋποθέσεις για τη θέση σε εμπορία των ε, δομικών προϊόν, προϊόντων κατασκευής Σύμφωνα με το άρθρο του κανονισμού εγκρίνεται αυτή η διόρθρωση. Πρόκειται για το άρθρο 216 παράγραφος 4. Ε, βεβαίως ε, εκτός ε, εάν σηκωθεί ο απαραίτητος αριθμός των βουλευτών για να ζητήσουν την άρση αυτής της διόρθωσης. Η δεύτερη ανακοίνωση με βάση το άρθρο 211 παράγραφος 3 Τη επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων προτείνει την εξή ερμηνεία των άρθρων 56 και 50. Ε, πρόκειται για την ερμηνεία του άρθρου 56. Με βάση την παραπομπή στην Επιτροπή και με βάση το άρθρο 56 παράγραφος 3 η αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας πριν αποφασίσει για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί ε, θέλει να επιτρέψει σε μια ε, αρμόδια επιτροπή να κάνει τις δικές επιλογές για τις τροπολογίες που είναι δική της αποκλειστική αρμοδιότητα κυρίως όσον αφορά την επιλογή των τροπολογιών που πρέπει να υποβληθούν εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η προθεσμία με βάση το άρθρο 3 δεύτερο κόμμα ε, και με βάση την προφορική πρόταση αφορά την αρμόδια επιτροπή. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να ορίσει την κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε να εξεταστεί η διαδικασία. Η ερμηνεία του άρθρου 50 και η απόφαση της διάσκεψης των Πρόεδρων να εφαρμοστεί η διαδικασία με τις συναρμόδιες επιτροπές αφορά όλη τη φάση της διαδικασίας και τα δικαιώματα της αρμόδιας επιτροπής ε, εφαρμόζονται από την ίδια την επιτροπή. Η εκτέλεση αυτών των ε, δικαιωμάτων βεβαίως και πρέπει όμως να σέβεται την αρμόδια επιτροπή και να τηρηθεί το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα. Το δικαίωμα τη ε, συναρμόντης επιτροπή είναι να καταθέσει τι ε, τροπολογίε. Και αυτό στο πλαίσιο των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων. Στην περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια επιτροπή επί της δεν αναγνωρίζει τι ε, πρόνοιε τη συναρμόντης επιτροπή, τότε οι αποφάσει που θα ληφθούν από την πρώτη παραμένουν ενισχύ. Όμω η συναρμόδια επιτροπή μπορεί να καταθέσει άμεσα στην Ολομέλεια τι τροπολογίε στο πλαίσιο των δικών τη των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων. Αυτή λοιπόν η ερμηνεία γίνεται αποδεκτή εκτός εάν υπάρχει αντίρρηση από την ε, ημερομηνία ένα των εργασιών που είναι αύριο ή Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτή την ερμηνεία τότε η έκθεση Ματιού θα αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη της ε, Ολομέλειας αυτής της εβδομάδας. Τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τις ε, ψηφοφορίες. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία με βάση την απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση «Ζολή» και για την ε, τροποποίηση, πρώτη τροποποίηση συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση Νοτιοαφρική για το εμπόριο, την άπτυξη και την συνεργασία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Θα ψηφίσουμε για αυτήν την έκθεση με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίθηκε η έκθεση. Η μερίσια διάταξη προβλέπει με την διαδικασία την ε, ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Κοπά που ε, αφορούν τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, Λιχτενστάν και της Νορβηγίας. Ψηφίζουμε λοιπόν για την έκθεση αυτή. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ε, λειτουργεί το μηχάνημα. Μπορείτε να στείλετε κάποιο τεχνικό. Κοφεράτη. Παρακαλώ κύριε Κοφεράτη. Και εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα. Δεν λειτουργεί ούτε η δική μου συσκευή. Παρακαλώ να καταγράψετε και τη δική μου την ψήφο. Ε, θα ληφθεί αυτό υπόψη από τι αρμόδιε υπηρεσίε. Τώρα λοιπόν η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφορία με την ίδια διαδικασία για την έκθεση